Good um, Καλό σας απόγευμα. Όπως είχα ανακοινώσει το πρωί θα αρχίσουμε κατευθείαν στις 3 η ώρα με το σημείο 16 που θα ακολουθηθεί από το 15 το 17 και μετά το 14. Ξεκινάμε τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά με εισηγητή τον Γιούργεν Κρόιτσμαν. Έχετε το λόγο κύριε Κρόιτσμαν για να ξεκινήσετε την ε, παρουσίαση της έκθεσης για τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση. Σας ευχαριστώ. Γερμανικά. Ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες οι οποίες οπωσδήποτε θα συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα της γνωμοδότησης. Τροπολογία 13 αναφέρει το σημαντικό ρόλο της Eurostat για την ελευθερία κίνησης, ε, κίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία ξεχωριστή παράγραφο. Και δεν ε, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Το ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση και όσον αφορά το θέμα εξέβρεσης απασχόλησης σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και όλα τα συναφή ζητήματα. Δυστυχώς ε, δεν ξέρουμε ακόμα. Ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι ακόμα πληροφορημένοι για όλο αυτό το πακέτο ενημέρωσης και γι' αυτό είναι πολύ καλό η Επιτροπή Απασχόλησης να προωθήσει ε, την ενημέρωση για την EURES. Εν συνεχεία αναφέρουμε στην κεντρική υπηρεσία παροχής πληροφοριών για όλα τα θέματα της ενιαίας αγοράς συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, των διατάξεων της εσωτερικής αγοράς για να μπορέσουν να προσεγγίσουν οι πολίτες πολύ καλύτερα ε, τους κανονισμούς αυτούς και να εκμεταλλευτούν όλες τις προσφορές που υπάρχουν και τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Ε, παρακολούθησα ημερίδες εργασία, σεμινάρια του Eurochamber και άλλων οργανισμών όπου αναφέρθηκε ότι οι ενδοκοινοτικές επαφές δεν έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά. Πολλές φορές αναφέρεται βέβαια μία υπηρεσία που μπορεί κανείς να αποτανθεί, καμιά φορά και σε άσχημα αγγλικά που δεν βοηθούν τους πολίτες μας. Λοιπόν, τι όφελος έχει όλη αυτή η δουλειά την οποία κάνουμε όταν δεν ενημερώνουμε τους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο ενημέρωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην παράγραφο 5 αναφέρουμε ότι πολλές αρμοδιότητες είναι εθνικές και ε, αυτές οι εθνικές αρμοδιότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν και να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν στις εθνικές υπηρεσίες όταν δεν λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση στο θέμα της ανάπτυξης των δικαιωμάτων των πολιτών για την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα ολίγα. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι. Τότε προ... Α, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αξιόλογο έργο σας. Έχω καταθέσει εξτροπολογίες η πιο σημαντική πιστεύω ότι είναι η παριθμό 16. Το θέμα της ε, της οικονομίας ακόμα εξακολουθεί να είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα ιδιαίτερα το θέμα της παραοικονομίας ή της γκρίζας, της φαιάς οικονομίας. Θα ήθελα η Κομισιό να μας δώσει κάποια απάντηση για τα θέματα αυτά, όπως είχε ζητήσει ήδη το Κοινοβούλιο το 2009. Επίσης θα θέλαμε να είχαμε σαφείς κανόνες ως προς τις υπεργολαβίες, γιατί όλο και περισσότερο οι υπεργολαβίες αυτές γίνονται διαμεθοριακά. Στη Φιλανδία, στη δική μου χώρα, κατασκευάζουμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο όπου υπάρχουν υπεργολάβοι από δεκάδες χωρών. Έχουμε και μια κυπριακή εταιρεία η οποία στέλνει Πολωνούς εργάτες οικοδομής στην Φιλανδία. Δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνο αν συμβεί κάτι όταν έχουμε μια μακρά αλυσίδα υπεργολάβων. Τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυτή την προβληματική και το τονίζω. Και η τροπολογία 17 επίσης, εναλλακτικές μέθοδοι ε, επίλυση διαφορών. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο στον τομέα των διαφορών που εμπλέκουν καταναλωτές. Θα ήταν όμως ενδιαφέρον να φέρουμε το θέμα αυτό και στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και διαφορών για να αποφύγουμε πολύ δάπανε και επαχθεί υποθέσει ενώπιον των δικαστηρίων. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο από την Κομισιόν να λάβει το λόγο στο σημείο αυτό. Είμαι η κυρία Μπρίντερ από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγοράς. Η ερώτησή σας για την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1 είναι αρμοδιότητα της Επιτρόπου κυρίας Ρέντιν και θα πρέπει να συζητήσω με τον συνάδελφό μου για θέματα δικαιοσύνης ε, και θα σας απαντήσω για αυτό το θέμα της αναθεώρησης που δεν το έχουμε χειριστεί ακόμα μέσα στο πλαίσιο της ε, ενιαίας αγοράς. Ε, η πρόεδρος, ο κύριος Κρότσμαν. Δεν θα σχολιάσω τις προτάσεις. σε αυτά που είπε η Φιλανδή συνάδελφος και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα στον ανταγωνισμό όταν π.χ. όπως είπε στο παράδειγμά σου στην Πολωνία εργάζονται εργάτες από την Κίνα με χαμηλότερους μισθούς. Η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή όσον αφορά το θέμα του δίκαιου και θεμητού ανταγωνισμού και η τροπολογία σας επιστεί την προσοχή σε αυτό το θέμα και δεν βλέπω πρόβλημα. Η 14 Φεβρουαρίου, λέει η Πρόεδρος, είναι η υιοθέτηση ε, στο Κοινοβούλιο και της γνωμοδότησης στις 2 Μαρτίου. 2 Μαρτίου θα ψηφιστεί. Θα υιοθετηθεί η γνωμοδότηση. Και Προχωρούμε στο 17 γιατί ο συγητής για το σημείο 15 δεν είναι εδώ. Προχωρούμε στο 17 λοιπόν και πάλι η κυρία Λίζα Γιακονσάρη που είναι η ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους και της δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έδειξαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τη γνωμοδότησή μου και υπέβαλαν συνολικά 80 τροπολογίες και πιστεύω πιστεύω ότι όλες αυτές τις τοπολογίες προσθέτουν πράγματι αξία στη γραμμοδότησή μου. Έχουμε τον ίδιο στόχο να εδραώσουμε σαφείς και αποτελεσματικούς στόχους ε, για την ενιαία αγορά ε, και, και σαφείς διατάξεις και ε, όλο αυτό το πακέτο έχει ως σκοπό να ωφελήσει τους πολίτες μας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποιοι είναι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδών, ε, οι επιχειρηματίες, οι πολίτες, τα παιδιά, ενήλικες. Έχει λοιπόν ένα πολύ ευρύ φάσμα ισχύω και γι' αυτό ακριβώς και τόσες τροπολογίες. Ε, βλέπω, διαβλέπω μέσα από όλες αυτές τις τροπολογίες ότι οι στόχοι μας παραμένουν κοινοί. Συνάδελφοι, κατανοώ ότι δεν έχουμε χρόνο να εξετάσουμε αναλυτικά όλες τις τροπολογίες. Οπότε θα αναφερθώ στα κέρια σημεία. Όπως είπα και νωρίτερα, Ε, ε, τα σημεία εκείνα που αφορούν υπηρεσίες, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Πιστεύουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα διότι είναι εξαιρετικά σημαντικές όπως η παροχή ε, νερού, ηλεκτρικού, η υποδομή η μεταφορική. Και ευχαριστώ τους κυρίους Κρότσμαν και Μπάλτασαρ όπως και την κυρία Πέρες για την τροπολογία 3 και πιστεύω ότι θα βρούμε ε, κατάλληλες λύσεις στη διατύπωση. Όλο το θέμα των υποδομών πραγματικά ε, πρέπει να το καλύψουμε σε μια ξεχωριστή παράγραφο, όπως προτείνει και η τροπολογία 33. Σύμφωνα και με, το, με τους κύριους Κρότσμαν και Μπάλτασάρ στην τροπολογία 17 ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τι ισχύει για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, ενδιαφέροντος SSGI. Και θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πιο σαφείς. Διαφορετικά θα δημιουργηθούν προβλήματα και θα βρεθούμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Γεγονός που δεν, το θέλουμε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Συζητήσαμε ήδη την κοινωνική ρήτρα και πιστεύουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να γίνουν σεβαστά σε όλες τις νομοθετικές πράξεις και στην τροπολογία 27 τη δικιά μου θέλω ακριβώς να διευκρινίσω αυτήν την αρχή και αναφέρω συγκεκριμένα το δικαίωμα της απεργίας και το, το δικαίωμα της διατήρησης και προστασίας δικαιωμάτων. Η ιδέα μου, η βασική μου ιδέα ήταν να υπάρξει μία ε, υποχρεωτική ρήτρα δεδομένου ότι αυτή η, ε, η ιδέα υποστηρίζεται από όλους τους συναδέλφους. Τροπολογία 24 από, τους, από τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ ε, συνδυάζεται, ε, αναφέρεται στην παράγραφο 9. στο άρθρο 9, συγγνώμη, των νομοθετικών προτάσεων, το άρθρο 9 της συνθήκης. Και επίσης είδε ενός ειδικού ε, δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι μια κακή ιδέα. Το έχουμε συζητήσει. Δεδομένου ότι στο Λουξεμβούργο εκδικάζονται πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις και υπουργό εργασία στη Φιλανδία όταν διατυπώνονταν αυτή η οδηγία I can see that... για την απόσπαση εργαζομένων και πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Βλέπω από τις ε, τροπολογίες ε, ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική πλέον και πρέπει να ε, κάνουν διάφορες αλλαγές. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η υλοποίηση και η εφαρμογή είναι ικανοποιητική αυτή τη ε, οδηγία. Άλλοι πιστεύουν το αντίθετο. Πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό αν θα την αναθεωρήσουμε ή όχι. Εν συνεχεία, τροπολογία 54. Κρότσμαν Μπάλτασα είναι εξαιρετικά καλή και σίγουρα θα βρούμε ένα συμβιβασμό είναι γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παίξουν έναν κέριο ρόλο στον ευρωπαϊκό μηχανισμό για τη βιομηχανική αναδιάφρωση και τέλος αυτή η επαγγελματική κάρτα που προτείνεται συμφωνώ ότι μπορούμε να, να συνδέσουμε την επαγγελματική κάρτα με το ε, διαβατήριο δεξιοτήτων, έτσι ώστε, όπως το λέμε, έτσι ώστε να υπάρχει μία κάρτα μόνο η οποία να περιλαμβάνει όλες αυτές τις πληροφορίες. Τροπολογία 65 είναι αυτό. Πιστεύω ότι αυτή η επαγγελματική ε, ε, κάρτα μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα και για εργαζόμενους και για εργοδότες. Πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο αυτό το θέμα, αυτή την πρόταση. Ε, και πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο στην ε, διευκόλυνση της λειτουργίας ε, της ενιαίας αγοράς. Και χαίρομαι που η Κομισιόν επιτέλους δέχτηκε να εξετάσει αυτό το, προτινόμενο, αυτό το θέμα της προτινόμενης εργασιακής ή επαγγελματικής κάρτας ταυτότητας. Και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους μου και τους κύριους Κρότσμαν και Μπάλτασαρ. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια κοινή διατύπωση, ένα συμβιβασμό που, ε, για, όλη τη γνωμοδότηση. Η πρόεδρος. Κάποιο θέλει να λάβει το λόγο ή κάποιο από την Κομισιόν ίσω θέλει να λάβει το λόγο, όχι. όχι. Σα ευχαριστώ τα μάλα. Η προθεσμία, μάλλον στι 14 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα θα εγκρίνουμε την ε, έκθεση αυτή στην Επιτροπή μας. Και, χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το υπαριθμό 15 για την εσωτερική αγορά. Ο κύριος ε, Μπαλτασάρη. Σα σας Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νιώθω ικανοποίηση μετά από τις 66 τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν στο σχέδιο έκθεσης στις περισσότερες περιπτώσεις, βελτιώνει το κείμενο και συμβάλλουν στους βασικούς στόχους που εξυπηρετεί αυτή η έκθεση. Δηλαδή, καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά, μειώνοντας το διοικητικό άχθος για αυτές τις επιχειρήσεις, διευκόλυνση των, της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίων, να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους διαγωνισμούς για να επιτευχθούν κοινωνικοί στόχοι και συντονισμός με τη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική. Στο φως αυτών των τεσσάρων στόχων συμμερίζομαι την αίτηση του, της κυρίας Όρονεν <clears throat> να υποστηρίξουμε τις ε, επιχειρήσεις που είναι ενεργές στον κοινωνικό τομέα, τροπολογίες 1 και 2. Συμφωνώ σε αυτό που είπαν διάφοροι συνάδελφοι για την κοινωνική διάσταση της ενεργείας αγοράς και την ανάγκη να έχουμε μία αηφόρο ανάπτυξη <clears throat> της ενιαίας αγοράς για να έχουμε θέσει εργασίας ποιότητος, όπως λέει η τροπολογία 6, η 14, η 18 που πάει. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ενιαίας αγοράς, ως ε, είπε ο κ. Κάμπροκ, στην τροπολογία 4, και φυσικά θα το συμπεριλάβω αυτό στην Συμβιβαστική τροπολογία. Δέχομαι θετικά τι τροπολογίες στην τρίτη παράγραφο σε σχέση με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην, ε, στη χρηματοδότηση με τις τροπολογίες Ράπτη και Κρόιτσμαν ζητούν συγκεκριμένες προτάσεις από, τα, από την πρόεδρό μας, την κυρία Μπερές. Νομίζω ότι στην πέμπτη παράγραφο όπου ζητείται συμπερίληψη κοινωνικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωση με τρίτες χώρε μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτές σε μια συμβαστική τροπολογία. Και στην τροπολογία 28 Κρόετσμαν, 21 Κονζούλη 31 Κρίστενσεν, 32 Γκαρζάλη. Θα προσπαθήσω να βρω μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ε, των κοινωνικών θεμάτων και την άρση των εμποδίων στο δημόσιο χώρο. Ούτω η τροπολογία 34 που πάκει είναι μια πολύ καλή βάση συμβασμού χάρη στην εκπεφρασμένη της μνήα της κοινωνικής υπευθυνότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στα πλαίσια της σύναψης εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Σημερίζομαι την αίτηση του κυρίου Ρένιερ σε σχέση με την ανάγκη να έχουμε ένα σωστό επίπεδο διαφάνειας, αυτή είναι η τροπολογία 40, για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των πιστωτών κατά τη διάρκεια των, ε, τροποποίηση της τροποποίησης των λογιστικών προτύπων, αλλά αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να μειώσει και το διοικητικό άκρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις απελευθερώσει από κάποιες απαιτήσει οι οποίες είναι πια πεπαλαιωμένες μέσα στο λογιστικό πλαίσιο και από την άποψη αυτή δεν θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κακώς εννοούμενη απορρίθμιση, όπως λέει η τροπολογία 38 της κυρίας του, Ρούνεν, ή, ή όπως λένε στην τροπολογία 39, 38 και 39 του Ρούνεν και Ράπτη, ότι θα έχει προβλήματα, θα δημιουργήσει προβλήματα για τους εργαζόμενους για την τροπολογία της κυρίας Σάρη, που θέλει να υπάρχει μια κοινή εδρεωμένη, παγιοποιημένη μάλλον ε, βάση φορολογίας των, ε, των επιχειρήσεων ώστε έτσι θα μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης με τεχνικά συστήματα φορολογίας και τέλος συμμερίζομαι απόλυτα την αίτηση της ε, Προέδρου Μπέρες στην τροπολογία της 55 για την πρόταση 17 και την νομοθεσία, το Single Market Act, την πράξη για την ε, ενιαία αγορά σε ό,τι αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και αυτό μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο, συστατικό στοιχείο της μιας συμβαστικής τροπολογίας γιατί αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα που είναι η πρόσβαση σε δημόσιους πόρους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να βελτιωθεί η καινοτομία, η κοινωνική συνοχή και η απασχόληση. Θα συντάξω προσφανώς για όλες τις παραγράφους όπου είναι δυνατόν τροπολογία συμβασμού. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο για το σημείο αυτό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό θέμα. Η παραδείγματο χάρη η τροπολογία 47 η δική μου αφορά τους φορολογικούς παραδείσους και εμείς το καταπολεμήσαμε αυτό και θα ήθελα να γίνουν περισσότερα από την Κομισιόν για να καταπολεμηθεί γιατί χρειαζόμαστε και κίνητρα και κυρώσεις διότι η φοροδιαφυγή, και οι παράνομες κινήσεις του κεφαλαίων είναι κάτι που το ταυτίσαμε από καιρό και το ζητήσαμε ήδη πέρυσι στα πλαίσια της καλής διακυβέρνησης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, μπορεί η Κομισιόν να μου πει τίποτε για το τι προτίθεται να κάνει για τους φορολογικούς παραδείσους, διότι μειώνεται η αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών άμα δεν πούμε ότι θα κάνουμε τίποτα. Απ' την άλλη, μήπως μπορείτε να μου ξαναπείτε όπως λέω στην τροπολογία 48 αυτός ο φόρος των δοσοληψιών των χρηματοπιστωτικών δοσοληψιών που ζήτησε το ΕΛΚ πέρυσι στην έκθεση Πρέπει να επαναληφθεί και εδώ, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Μήπως κανείς άλλος. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια νέα βάση υπολογισμού φόρων. Αυτό θα βοηθούσε πολύ και δυστυχώ δεν έχουμε αυτή την ενιαία βάση. Γι' αυτό, εφόσον δεν, το, δεν έχουμε αυτή την κοινή βάση, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το φορολογικό ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να το καλύψουμε το ΦΠΑ, την έλλειψη αυτής της βάσης, διότι, εάν θέλουμε, να βοηθήσουμε ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν είχαν ΦΠΑ ε, 10% μετά ξέσπασε η κρίση μέσω, με τη βοήθεια της Ιρλανδίας και των χαμηλών φορολογικών συντελεστών η οποία η Ιρλανδία προσέλκυσε πάρα πολλές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ε, χαμηλή, τους χαμηλούς φόρους ε, αλλά ε, αφόσον δεν έχουμε νέα φορολογική βάση, νέο φορολογικό συντελεστή, ας πούμε ότι θα θέσουμε ένα μήνυμο επίπεδο για λόγους αλληλεγγύης. Ε, τα υπόλοιπα θα διαχειριστούν τα κράτη-μέλη. Έχουμε κράτη τα οποία έχουν υψηλότερο συντελεστή βασικής φορολογίας και άλλα κράτη με χαμηλότερο συντελεστή βασικής φορολογίας. Ας το αφήσουμε αυτό έτσι. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κοινωνικά συστήματα σε ορισμένες χώρες που χρηματοδοτούν χρηματοδοτούνται από τους φόρους. Αλλά κοινωνικά συστήματα όπως η Γερμανία χρηματοδοτούνται από εισφορές, δεν, κοινωνικές εισφορές. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καθιερώσουμε έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή. Ο ανταγωνισμός είναι σωστός εφόσον είναι θεμητός. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ενιαία βάση υπολογισμού ξεκινώντας επί τη βάση ενιαίου ε, ενιαίας, ενιαίου τύπου υπολογισμού ήδη θα έχουμε επιτύχει πρόοδο. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Μπαλτασάρ, Μπαλτασάρε, Έχουμε 28 από εμά έχουμε ζητήσει, α, στην τροπολογία 28 ζητιέται η συμπερίληψη διεθνών προτύπων στις εμπορικές συναλλαγές. Βεβαίως ε, πιστεύω ότι η συμπερίληψη προτύπων ε, άλλων τρίτων χωρών μπορεί να είναι μια καλή ιδέα, αλλά δεν μας ωφελεί εδώ. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κοινωνικά πρότυπα σε εμπορικέ συμφωνίες ε, όπου είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτά, ε, διότι είναι προς το συμφέρον μας αυτήν την τροπολογία 28 που έχω υποβάλει. Έχουμε επίσης υποβάλει μια τροπολογία για τα βιομηχανικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε τα πνευματικά δικαιώματα διότι αποτελούν ε, ε, τμήμα της νομοθεσίας μας ε, διότι αυτοί οι οποίες συμβάλλουν δημιουργούν και πνευματικό προϊόν το οποίο συμφέρει και προωθεί την κοινωνία και γι' αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν είναι δυνατόν τα δικαιώματά τους να χάνονται ή να μην τα λαμβάνουν λόγω ίντερνετ, διαδικτύου και άλλων τεχνικών μέσων. Η, η πρόεδρος, η Κομισιόν θέλει να παρέμβει, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώς να υπογραμμίσω τη σημασία του να υπάρχει μια κοινωνική ρήτρα στις εμπορικές συμφωνίες. Όπως ξέρετε, σε μια πρόσφατη ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ευρώπη έχουμε αναφέρει πια είναι η πολιτική μας για τα θέματα αυτά και η Κομισιόν προσπαθεί πάντα να διαπραγματεύεται τη συμπερίληψη τέτοιων προτύπων ρητρών σε διεθνείς συμφωνίες και αυτό συμπεριλαμβάνει και τις διμερείς συμφωνίες. Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο όλες οι συμφωνίες να εξασφαλίσουν τη συμπερίληψη μιας τέτοιας ρήτρας, ιδίως αν είναι πάρα πολύ ειδικέ και με περιορισμένη εμβέλεια. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό το οποίο είπε ο κ. Κρόισμαν, πρέπει να έχουμε ευελιξία στο σημείο αυτό, αλλά η βασική πολιτική της Κομισιόν είναι πράγματα συμπεριλαμβάνονται τέτοιες ρήτρες. Γυρίζω στον κύριο Μπαλτασάρη για να κάνει την σύνοψη την τελική. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπαλτασάρη. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Οι δύο τροπολογίες οι οποίες αναφέρθηκαν από την κυρία Γιακονσάρη για τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν έχουμε την ίδια εμπειρία όλες τις χώρες μας φυγής κεφαλαίων προς ε, φορολογικούς ε, παραδείσους όπου οι πόροι αυτοί οι οποίοι θα ήταν πολύ χρήσιμοι για την ευρωπαϊκή οικονομία χάνονται. Δεν νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότησή μου είναι ο κατάλληλος χώρος, ο πιο, ο εύστοχος χώρος για να κάνουμε αυτήν την προβληματική και να διατυπώσουμε το αίτημα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη και πιο σωστή αντιμετώπιση της αντιμετώπισης του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων. Η τροπολογία φυσικά είναι τεκμηριωμένη, αλλά είναι λιγάκι εκτός παιδιάς σε σχέση με το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Αντίθετα, η 48, η οποία ζητά την ε, επιβολή ενός φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, έχει ήδη διατυπωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο σχετικά έχει ζητήσει μονάχα να εκπονηθεί μια μελέτη σχετικά. Ενώ αντίθετα η πρόταση που πολλέ φορέ η ίδια η πρόταση για τον φόρο έχει προσκρούσει πολλέ φορέ σε άρνηση του Συμβουλίου Υπουργών γιατί υπάρχει στεναρή αντίδυση ορισμένων κρατών να εφαρμοστεί ένας φόρος στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Μου φαίνεται λοιπόν περιττό και άσκοπο να το προτείνω αυτό και πάλι σε μια έκθεση η οποία δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να δοκιμήσει το σενάριο μιας ε, φορολογίας τη στιγμή που ξέρουμε ότι το Συμβουλίο δεν θα δεχτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Από ό,τι ξέρουμε τώρα, δεν υπάρχει καμία συνένεση στο Συμβούλιο για ένα τέτοιο φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Συμφωνώ προφανώς ότι είναι απαραίτητο το φορολογικό σύστημα να έχει κάποιο κοινό γνώμονα. Είναι μια άποψη την οποία Μπορούμε να τη δεχτούμε πιστεύω όλοι. Και ουσιαστικά είναι οξύμορο να έχουμε ενιαίο νόμισμα και συγχρόνως να έχουμε εθνικούς προϋπολογισμούς, διαφορετικά συνταξιοδοτικά πλαίσια και διαφορετική φορολογική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό και πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να προσπαθήσει να δημιουργήσει και κοινέ βάσεις, αλλιώς όπως έχουμε δει ήδη θα εξακολουθεί να, να διατηρείται μια κατάσταση η οποία δεν στέκεται. Δεν μπορεί σε κάποιες χώρες να συνταξιοδοτείται κάποιο στα 68 και αλλού στα 50 ή σε άλλες χώρες να είναι πολύ λίγοι πολίτες οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 100.000 ευρώ το χρόνο και την ύφη την πληρώνουν άλλοι πολίτες που έχουν πολύ χαμηλότερο εισόδημα και αυτό οδηγεί σε ένα τεράστιο δημόσιο χρέο. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει <clears throat> ένα κοινό νόμισμα το οποίο καλύπτει 16-17 χώρε μα. Πρέπει λοιπόν επίση και για την ε, πνευματική διοκτησία να εξασφαλίσουμε την ε, προστασία τη πνευματική διοκτησία, κάτι που καλύπτεται ήδη από ορισμένε οδηγίε. Και η συμβαστική τροπολογία που δεσμεύομαι να σας φέρω, προφανώς θα, λάψει, θα λάβει υπόψη το πρότυπο αυτό των <clears throat> κοινωνικών, των κοινών κοινωνικών προδιαγραφών και πιστεύω ότι θα πρέπει να το εφαρμόσουμε αυτό με στεναρότητα αλλά και με την απαραίτητη ευελιξία δεδομένου ότι στις διεθνές σχέσεις <clears throat> υπάρχουν χώρες που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να τις σεβαστούμε αν θέλουμε να έχουμε συμφωνίες μαζί τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφής η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν να σεβαστούμε τα κοινωνικά πρότυπα, να δώσουμε κίνητρα στα κοινωνικά πρότυπα, αλλά πάντα με την απαραίτητη ευελιξία. Για να συνεχίσουν οι εμπορικές ροές, οι οποίες είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου Στρασβούργο και στο, στην Ολομέλεια 2 Μαρτίου. Και τέλος το σημείο 14 Εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής η προώθηση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δίνω το λόγο στον κύριο Φάλμπρο, συγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έκθεση ε, είναι πολύ επικριτική στο το ύφος της, διότι σε πολλά σημεία της έκθεσης αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική της διάσταση πολλές φορές δεν έχει μία συνεπή συμπεριφορά. Πολλές φορές μάλιστα είναι υποκριτική ενώ προσπαθούμε να είμαστε μοντέλο, πρότυπο για τις άλλες χώρες του κόσμου, ε, άρα θα πρέπει να συμπεριφερθούμε και ανάλογα. Σε, με πολλές χώρες έχουμε εμπορικές συναλλαγές και τους ζητούμε να συμπεριφέρονται ευπρεπώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και εμείς ανάλογα, με συνέπεια και ευπρέπεια. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα αυτό έχει ε, οδηγήσει σε καυτές, έχουν γίνει καυτές θερμές συζητήσεις επί του θέματος αυτού ε, και λέμε λοιπόν ότι ε, η γυναίκα του Κέστρα πρέπει να, όχι μόνο να φαίνεται αλλά και να είναι όχι μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται τίμια στην περίπτωση της Τινησίας βλέπετε που έχουμε φτάσει. Έχουμε μία συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την χώρα αυτή, με την Τινησία. Άρα λοιπόν θεωρητικά θα πρέπει η χώρα αυτή να σέβεται τα ίδια πρότυπα, τα ίδια στάνταρτ. Τώρα βέβαια ξέρουμε τι έχει γίνει στην Τινησία το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Ας μην σήξουμε την Αίγυπτο. Ακούμε για κοινωνικό διάλογο, την, το σεβασμό ε, ε, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Υιοθετούμε και συμφωνούμε επί εκατοντάδων κειμένων, τα οποία μετά ξεχνάμε, επί της ουσίας ξεχνάμε. Τι δεχτήκαμε, τι ψηφίσαμε. Όσον αφορά δε, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ξέρουμε ότι η επιρροή του ΔΟΕ έχει μειωθεί και η ισχύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εργαζομένων και αυτή φθήνει μέσα στα πλαίσια του ΔΟΕ. Υιοθετήσαμε επίση ένα σχέδιο ε, Έχουμε συζητήσει ένα σχέδιο οδηγία το οποίο είναι αντίθετο στι αρχέ του ΔΟΕ. Και η Λισαβόνα και η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 αναφέρεται επιμακρών σε κοινωνικά θέματα και στην κοινωνική διάσταση, όμως στην πραγματικότητα επικεντρώνεται περισσότερο στον ανταγωνισμό. Και ε, όμως είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική πάση θυσία. Οι βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, σέβονται ταυτόχρονα και τον κοινωνικό διάλογο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτό πράγματι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η συνεργασία. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου θα έχουν πολλά να παρατηρήσουν, πολλά να πούνε στη συζήτηση αυτή. Δεν περιμένω πολλές τροπολογίες ε, ή μάλλον διορθώνω αυτό που είπα, δεν θα ήμουν ευτυχής εάν δω να υποβάλλονται πολλές τροπολογίες, διότι αυτό σημαίνει αποδυνάμωση της γνωμοδότησης και αποδυνάμωση της αρχικής θέσης του εισηγητή. Ας πω τώρα μερικά μόνο πράγματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν υπάρχει πια η διασύνδεση μεταξύ ε, μιας εταιρείας και μιας συγκεκριμένη τοποθεσίας όπου εδρεύει αυτή η επιχείρηση. Όταν μιλάμε για εταιρική κοινωνική ευθύνη, μιλάμε για μια ε, υπερεθνική διασυνοριακή ευθύνη, διότι μια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της ή μέσω ενός δικτύου θηγατρικών να λειτουργεί σε πολλές χώρες κλπ. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να επιδιώκουμε για την εταιρική ευθύνη κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Είμαι πρώην συνδικαλιστής και αναγνωρίζω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν υπονομευθεί. Όπως σας είπα, η επιρροή τους ε, αποδυναμώνεται και παρόλο που συνεχώς αναφερόμαστε στο σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, στον κοινωνικό διάλογο, βλέπουμε μία αποδυνάμωση αυτών των στοιχείων. Αναφέρουμε στη γνωμοδότησή μου επίσης ε, τα, δικαιώματα, ε, τα, τα, δικαιώματα σε βιομηχανικούς και σε πε, πε, ζώνες, σε ε, μετακινούμενους εργαζόμενους και ζητώ τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Όμως αυτό τελικά που βλέπουμε να γίνεται είναι μια, ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι ε, στην εργασία τους υποβασμίζονται όλο και περισσότερο κακής ποιότητας εργασίας και κακές συνθήκες εργασίας. Ε, όταν λοιπόν επιδιώκουμε βελτίωση των συνθήκων και των προτύπων στη, στο εσωτερικό μας πρέπει να το ζητούμε και από τους ε, εταίρους μας. Και πολλές φορές αναφέρονται στους κανονισμούς του ΠΟΕ. Πριν από μερικά χρόνια, όταν διαπραγματευόμασταν τον κανονισμό του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμποριού, Στη Σιγκαπούρη είχαν προσπαθήσει ορισμένες χώρες να προωθήσουν μια σκληρή σύμβαση επί της οποίας ε, θα λειτουργούσε ο ΠΟΕ. Τώρα όμως ε, ε, ξέρουμε βάσει των προτύπων του ΔΟΕ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Τώρα όμως ξέρουμε πόσο λαμβάνουν υπόψη τους τη ΔΟΕ. Ε, πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή θα δεχτεί την άποψή μου και τις παρατηρήσεις μου στο σχέδιο γνωμοδότησης και θα συμβαδίσει μαζί μου και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Διευθυντή της European Trading Foundation. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας που μου δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρω και εγώ στη συζήτησή σας. Ε, πολύ ταπεινά θα ήθελα να σας πω ότι την έκθεση αυτή τη θεωρούμε πολύ σημαντική γιατί η δουλειά μας γίνεται κυρίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμβαλόμενες χώρες, με εταίρους και η έκθεση μας δίνει μια πολιτική βάση στην εργασία μας. Ένα πολιτικό πλαίσιο μάλλον. Θα ήθελα για να σας πληροφορήσω για όσα αγνοείτε ως προς τη δική μας εργασία να πω σύντομα με ποιον συνεργαζόμαστε και μετά αν έχετε προτάσεις να κάνετε ευχαρίστως να τις ακούσω η μεταφορά και εφαρμογή του εγγράφου αυτού θα γινόταν με τα χαράς δεκτή από μας. Οι περισσότερες μας χώρες, 27 από τις 30 με τις οποίες συνεργαζόμαστε, είναι χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και η, κατα... η μείωση της ανέχειας αυτές είναι ουσιώδης. και οι χώρες και τα κόμματα καθώς και το ΓΑΜΑ 20 πρόσφατα στην εκπαιδευτική και μετεκπαιδευτική πολιτική είπε ότι όπως λέει και αυτή η έκθεση πολλές φορές πρέπει να υπάρξει στήριξη και προώθηση των δεξιοτήτων που διαθέτει το εργατικό δυναμικό εμείς εδώ δεχόμαστε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και ιδιαίτερα την επαγγελματική εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων διότι είναι βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανέχειας αυσές στις χαμηλοεισοδηματικές χώρες. Πρέπει λοιπόν στην εκπαίδευση μετά τη δευτεροβάθμια να αυξηθούν οι δεξιότητες, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού δεν έχει τη δυνατότητα να μείνει στην, ε, στον κύκλο της παιδείας μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο. Επομένως, για μας το σημαντικότερο είναι η σύνδεση μεταξύ παιδείας και απασχόλησης σχολείου και επιχειρήσεων. Γι' αυτό, επίσης, η στήριξη προς τις χώρες αυτές δεν θα συνίστατο μόνον στην καλή ποιότητα της παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είτε μιλάμε για νέους είτε για νεότερους, είτε για παιδες, αλλά και σε παιδεία και εκπαίδευση που να έχει σχέση με την επαγγελματική καριέρα, αν θέλουμε να μειωθεί η ανέχεια στις χώρες αυτές. Ακόμη σημαντικότερο στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι το θέμα της ανεργίας των νέων που αυξάνεται συνεχώς και όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από την κρίση και μετά. Και άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στην παιδεία και στην απασχόληση μειονεκτουσών ομάδων. Εδώ η δουλειά μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα της συνεργασίας που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των διάφορων κόσμων, όχι μόνο παιδείας και επιχειρήσεων, αλλά και του κόσμου της υποχρεωτικής εγκυκλίου παιδείας με την επαγγελματική τη αυτή. Εδώ πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό σε όλες τις χώρες και συντονισμός της κοινωνικής πολιτικής. Η έκθεση αυτή επίσης αναφέρεται στο εμπόριο. Πράγματι Πολλές εμπορικές συμφωνίες και συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ Ένωσης και δικών μας χωρών. Οι πρόσφατοι αριθμοί από τον ΠΟΕ δείχνουν ότι υπάρχει μία αλλαγή στις ροές του εμπορίου και οι περισσότερες ροές προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό χρειάζεται μια προσαρμογή για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ώστε οι απασχολούμενοι με το εμπόριο να ορίσουν ακριβώς που πρέπει να απευθύνουν τα εμπορεύματα προϊόντα και πού τις δεξιότητες των. Επίσης θεωρούμε ότι η ευθύνη των επιχειρήσεων είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να το καταλάβουν οι πολυεθνικές της Ευρώπης που εργάζονται ή δρούν στις χώρες μας, διότι είναι προφανές ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, στις επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν το θέμα και μερικοί από αυτούς θεωρούν ότι η επιχειρησιακή ευθύνη είναι πολυτέλεια, ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι το ουσιώδες και βασικό. Χαιρετίζουμε λοιπόν την αναφορά που γίνεται εδώ στην κοινωνική ευθύνη ιδιαίτερα διότι και οι δεξιότητες είναι τμήμα αυτής της ιδέας της ανάπτυξης μεγαλύτερης ευθύνης. Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά στην έκθεση αυτή από τις δικές μας απόψεως, από την άποψη δηλαδή των χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μπορέσουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες στις χώρες αυτές να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία αυτά βελτίωσης αν θέλουμε οι χώρες αυτές να προοδεύσουν. Είναι πολύ σημαντικό να λύσουμε τα προβλήματα και τα θεσμικά αλλά και τα θέματα της κοινωνικής εταιρικότητος. Οι εκπρόσωποι, οι εμπορικοί εκπρόσωποι της Ένωσης στις χώρες αυτές αλλά και άλλοι από την κοινωνία των πολιτών χρειάζονται αξιόπιστους εταίρους για τη συνομιλία και τη συνεργασία τους. Είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Για το 11 έχουν ήδη προγραμματιστεί οι δραστηριότητες μας, αλλά πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα είναι πολύ σημαντικά για μας. Προσθέτω κάτι μια διάσταση που ίσως να σας βοηθήσει για τη μετανάστευση ιδιαίτερα στις νότιες χώρες όπου συμβαίνουν πολλά ατυχήματα σε σχέση με τη μετανάστευση και προβλήματα σημειώνονται. Στις δικές μας χώρες προέλευσης πρέπει να γίνει η προσπάθεια ώστε μερικοί από αυτούς τους παράνομους μετανάστες να επιστρέψουν αλλά και οι νόμιμοι μετανάστες ή και εκείνοι που εθελοντικά επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την τυχόν εμπειρία τους για να αρχίσουν επιχειρήσεις και να βρουν κάποια δουλειά. Όλα αυτά συμφωνούν με τη συζήτηση που γίνεται τώρα στο ΓΑΜΑ 20 ως συνέχεια της Σεούλ. με συμμετοχή των εκπροσώπων της UNESCO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ΣΕΝΤΕΦΟΠ και του ΟΣΑ. Όχι του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, του ΟΣΑ. Όλοι αυτοί προσπαθούν να συνεργαστούν για να δουν ποιες δεξιότητες χρειάζονται περισσότερο οι χώρες χαμηλών εισοδημάτων και ψάχνουν επίσης στρατηγική που να είναι σε θέση να, να λύσει τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν. Η Ευρώπη νομίζω καιρό είναι πια να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να εκμεταλλευτεί την εμπειρία που έχει προς όφελος και άλλων χωρών για να μπορέσουν και αυτές να πάρουν μαθήματα από το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράς από την Κομισιόν, παρακαλώ. Όχι, δεν θέλετε. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Ή... Ή... Ο κύριος Σέρκος. Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την αναγνώρισή μου για το έργο του κυρίου Φάλμπρο γιατί αρκεί να βλεφαριάσει λίγα και κανεί την έκθεση για να δει το πόσο τεκμηρίωση υπάρχει πίσω τη, με πόση αυστηρότητα έχει συλλέξει τα στοιχεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά φυσικά είναι ιδιαίτερα πεπλεγμένα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο ίδιος, <clears throat> έχουμε ενώπιόν μας ένα στοιχείο που θα παίξει μεγάλο ρόλο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιμετωπίζουμε, κυρία Πρόεδρε, τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρήσαμε να διατηρήσουμε το δικό μας υπόδειγμα ζωής και εργασίας που κράτησε πάνω από ένα αιώνα με το να έχουμε ένα κοινό εγχείρημα αξιών που βασίζεται στην ε, αξιοπρέπεια των ατόμων και των εργαζομένων. <clears throat> Αλλά αντιμετωπίσαμε μια πραγματική επανάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι μια επανάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι νέος τρόπος παραγωγής, νέος τρόπος αγοράς και κατανάλωσης <clears throat> και επομένως βρίσκεται υπό αφισβήτηση και η ίδια η ευρωπαϊκή διάσταση σε τέτοιο σημείο που να πιστεύω ότι οι επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας για την επόμενη δεκαετία είναι ομές. Ή θα βρούμε αρκετά επιχειρήματα και αρκετή δύναμη για να δεχτεί ο κόσμος και να εργαστεί υπέρ ενός συστήματος αξιών όπως αυτό που έχουμε οικοδομήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας τρόπος εργασίας, διαβίωσης, μια σειρά από κοινωνικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή αλλιώς θα πρέπει εμείς να μιμηθούμε όλες αυτές τις άλλες χώρες που οι εργαζόμενοι ζουν στην επισφάλεια, στην έλλειψη δικαιωμάτων κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η επιλογή που έχουμε ενώπιόν μας. Θα πρέπει, θα πρέπει ή με, το παράδειγμά μας να κάνουμε τον κόσμο να προχωρήσει προς τα ή θα υπαναχωρήσουμε και εμείς σε εποχές όταν δεν υπήρχαν αυτά τα δικαιώματα όπως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε, στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου που μας ανταγωνίζονται σε μια αποκοσμιοποιημένη αγορά και οικονομία. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση μας και θέλω να πω στον κύριο Φάλμπρα ότι όπως και ο ίδιος <clears throat> συμφωνώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση κατεπίγουσας ανάγκης με πολλά προβλήματα γιατί έχουμε πολλή ρητορική η οποία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα του πρότεινα το εξή, ακόμα και αν είναι χειρότερα τα πράγματα, αν φτάνουν στο κόκαλο οι αντιφάσεις μας, θα πρέπει να πω ότι ίσως <clears throat> είναι υπερβολικά απεσιοδοξο ο κ. Φάλμπερ. Δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Εμείς ως Κοινοβούλιο που υποστηρίζουμε την κοινωνική Ευρώπη έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να πούμε και δεν πρέπει να έχουμε μια στάση παθητική απεσιοδοξίας είπε ένας Ισπανός φιλόσοφος ότι η γνώση και η σκέψη μας φέρνει πολλές φορές στην απεσιοδοξία, αλλά η θέλησή μας μας φέρνουν σε μια πιο αισιόδοξη αντιμετώπιση. Μια τελευταία παρατήρηση. <clears throat> Διάβασα ένα πολύ σημαντικό πόνημα πρόσφατα σε σχέση με τις συμφωνίες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που, και ιδιαίτερα στο, τη Συμφωνία Υπαριθμών 49 που είχε να κάνει με την περίπτωση Γκρούφε και τα προβλήματα με τις συλλογικέ συμβάσεις στην Γερμανία. Θα δώσω το κείμενο αυτό στον κύριο Φάλμπρετ, αυτή την πανεπιστημιακή διατριβή. Αυτό το οποίο μας διδάσκει αυτό το έργο είναι ότι <clears throat> η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον η ανάγνωση που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ανάγνωση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, η σύγκρουση μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει αποτέλεσμα όχι μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πιέζει τα κράτη-μέλη για να προσυπογράψουν τη σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αλλά αντίθετα τα κράτη-μέλη που έχουν δεχθεί τη Σύμβαση 94 να την αποκηρύξουν γιατί είναι ασύμβατη με την ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία διακίνησης των εργαζομένων και την απόσπαση εργαζομένων κτλ. Υπάρχουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία απέστησαν την υπογραφή τους από τη Σύμβαση Παριθμών 94 γιατί φαίνεται ότι θεωρούν ότι είναι κάτι <clears throat> το αντιφατικό με την ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια προβλήματα έχουμε να κάνουμε την οδηγία περί αποσπάσεως εργαζομένων και άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Εκεί θα καθοριστεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πω στον κύριο Φάλμπορ ότι θα ετοιμάσω και μια τροπολογία, όχι για να αυξήσω την ε, απεσιοδοξία του, αλλά για να δείξω την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Μια τροπολογία που να λέει ότι στην τελευταία κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιτροπή είχε δεσμευτεί για αυτό το οποίο λέει ο κ. Φάλμπερ στην έκθεσή του. Ότι να πιέσει τα κρατημέρια για να κυρώσουν τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Μία τροπολογία λοιπόν θα καταθέσω για να υπενθυμίσω αυτό το οποίο ξέχασε η Κομισιόν <clears throat> ότι υπάρχει υποχρέωση να πιέσει τα κράτη-μέλη να δεχτούν τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και να κυρώσουν αυτό το, αυτή τη σύμβαση γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο μόνο με το ηθικό μας ανάστημα ώστε να είναι σαφές ότι η Ευρώπη όχι μονάχα δίνει κηρύγματα προς τους άλλους, αλλά τηρεί και αυτά τα οποία κηρύσσει Ευχαριστώ. Κύριο Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω μερικές από τις σημαντικές αναφορές που ο Ρίκαρτ Φάλμπρο ανέφερε για το κείμενο αυτό. Καταρχήν, ο σεβασμός των κοινωνικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού υποδείγματος. Αυτό μπορεί να διατρέξει πάρα πολλές ενέργειες και δράσεις. Ήταν ιστορικά πάρα πολύ σημαντικά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Ήταν και ένα σημείο αναφοράς για την ταυτότητα εκατομμυρίων εργαζομένων και επέτρεψε στην Ευρώπη να αναπτυχθεί οικονομικά και να δώσει μια ιδιαίτερη σημασία στην εργασία και στους εργαζομένους σήμερα τίθεται ένα αμφιβόλο αυτό το υπόδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί υπάρχουν πια εταιρείε οι οποίες παράγουν και αγαθά και υπηρεσίες, αλλά θέλουν να εισαγάγουν συστήματα μέσα στα οποία τα δικαιώματα των ατόμων και τα κοινωνικά τους δικαιώματα παίρνουν άλλη διάσταση, μάλλον μειώνεται η διάστασή τους γιατί είναι πηγή πρόσθετου κόστους. Με την αλόγιστη λοιπόν αυτή προσπάθεια συμπίεσης του κόστους, <clears throat> στοιχεία που ήταν πολύ σημαντικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την ταυτότητά τους βρίσκονται υπό επίθεση. <clears throat> Έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον αλλά και λόγους πολιτιστικούς και πολιτικούς να υπεραμεινθούμε αυτού του υποδείγματος του ευρωπαϊκού του μοντέλου. Και η κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Υπήρου και των χωρών της ήταν και στο παρελθόν και τώρα ακόμα ένας λόγος προσέλκυσης επενδύσεων που επέτρεψαν στο μεταποιητικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί περισσότερο. Πιστεύω λοιπόν ότι η περάσπιση αυτού του μοντέλου και ε, εξάλλου που περιλαμβάνεται και σε πολλές συμφωνίες που έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, θα πρέπει να ισχύει και σε εμπορικές συμφωνίες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί συμφωνίες εμπορικές με χώρες όπου είναι φανερό ότι κατά συρροή λόγω ελλείψεως δημοκρατίας ή λόγω διαφορετικής προσέγγισης παραβιάζονται και τα κοινωνικά δικαιώματα και τα απλά ανθρώπινα δικαιώματα πολλέ φορέ των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται εκεί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Ρίκαρτ Φάλμπρο. Θα πρέπει να τονίσουμε <clears throat> την ανάγκη να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Δεν πρέπει να αποσύσουμε την δυνατότητα να, εμποδίσουμε τις εμπορικές ροές. Δηλαδή ότι μπορεί και εμείς να εμποδίσουμε την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται κάτω από συνθήκες που μας φαίνονται απαράδεκτες. Ένα δεύτερο σημείο είναι αυτό της κοινωνικής ευθύνης των εταιριών. Το εργαλείο της εταιρική ευθύνης είναι ένα κατά κάποιο τρόπο αμφίσιμο εργαλείο. Έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς και από πολλές εταιρείε σαν ένα στοιχείο προπαγάνδας. Προπαγάνδας, γιατί θεώρησαν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να περιγράψουν τις δραστηριότητές τους ως σεβόμενες το περιβάλλον, οδηγούσε σε ανάπτυξη ανθρώπινη. Πολλές λοιπόν πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες συγχρόνως ρίπαιναν της θάλασσα στη Βόρεια Ευρώπη και οι οποίες ε, φέρνανε πρώτες ύλες από πάρα πολύ μακριά και όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν επομένως να βγει αυτή η αρνητική πτυχή που έχει η εταιρική ευθύνη, ο καθαρά προπαγανδιστικός της χαρακτήρας και να περάσουμε από μια εθελοντική προσφυγή στην εταιρική ευθύνη σε μια δεσμευτική ρύθμιση όπως με μια οδηγία. Δεν μπορεί να είναι μονάχα θέμα image και αξιοπιστίας και φήμης μιας επιχειρήσεως που θα τις οδηγήσει να έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί την παιδική εργασία σε, στον τρίτο κόσμο και όταν έγινε αυτό γνωστό υπέσταν και εμπορικές ζημίες γιατί οι καταναλωτές έπαψαν να αγοράζουν τα προϊόντα τους. Αλλά αν είναι μονάχα εθελοντική αυτή η εταιρική ευθύνη θα έχουμε και στρεβλώσεις ανταγωνισμού θα υπάρξουν επιχειρήσεις που εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν ως φενάκι την εμπορική, την ε, εταιρική μάλλον ευθύνη, χωρίς να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα η οποία να εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία της εταιρική ευθύνη θα πρέπει να γίνουν εργαλείο, να δεσμευτικά και να δεσμεύουν όλες τις επιχειρήσεις. Να υπάρχουν λοιπόν μια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά εν καιρό και διεθνή πρότυπα. Η Πρόεδρος, η Κομισιόν είναι παρούσα, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μοράζ που ήρθε τώρα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που άρχισα. Πρόσφατα ακούσαμε για αυτές τις αλλαγές των σημείων της μερίστε διάταξης. Θα ήθελα να κάνω ε, μερικά σχόλια για την εξωτερική διάσταση. Ασφαλώς έχουμε δει μία πολύ ισχυρή έμφαση να δίνεται στην Ευρώπη και παγκοσμίως σε αυτά τα θέματα και αυτή, αυτές, αυτή η διάσταση, αυτή αυτή η δυναμική κίνηση θα πρέπει να διατηρηθεί για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ανάκαμψη με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των εξελίξεων είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να ασχολείται με το θέμα της εξωτερικής διάστασης, με το ψήφισμα που συζητιέται σήμερα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, διεθνή, στο τι γίνεται διεθνώς και τι συζητιέται διεθνώς στο πλαίσιο των G20 ε, και γενικά για την προσπάθεια ανάκαμψης σε παγκόσμια κλίμακα ε, ήδη η διεθνή Οργάνωση Εργασίας έχει προσπαθήσει να βοηθήσει σημαντικά την διεθνή ανάκαμψη και η Κομισιόν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα συνδράμει και εκείνη ε, βεβαίως πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς ε, και τις διατάξεις ε, του, του ΔΟΕ για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις κλπ. Θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη έχουν επιχειρώσει ε, τις ε, συμβάσεις ε, που αφορούν την εργασία του, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. όλες οι χώρες λοιπόν έτσι έχουν επικυρώσει και επίσης το θέμα της προστασίας των εργαζομένων. Ε, αυτό θα είναι και το βασικό θέμα των εργασιών της Γαλλίας ε, τον Ιούνιο. Η Κομισιόν δεν δραστηριοποιείται μόνο στη διεθνή, στο διεθνές επίπεδο, αλλά προσπαθεί επίσης να προωθήσει τον διάλογο με όλους τους στρατηγικούς εταίρους σε κοινωνικά και εργασιακά θέματα. Επίσης η Κομισιόν έχει συμβάλει επικοδομητικά στην πρόθεση αυτών των ζητημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Σας υπενθυμίζω ε, την Υπουργική Διάσκεψη του ΑΣΕΜ για ε, θέματα εργασιακά ε, στην περιοχή της ε, Μεσογείου που έγινε πέρσι, τον χρόνο της Λεκάνης Μεσογείου. Αυτή η εταιρική κοινωνική ευθύνη ε, έχει επιπτώσεις και σε άλλες πτυχές της πολιτικής, ε, ιδίως στην εμπορική πολιτική, στην πολιτική εμπορικών συναλλαγών. Γι' αυτό και η Κομισιόν θα προτείνει νέες, ναι, θα κάνει νέες προτάσεις σήμερα όσον αφορά ε, την μεθοδολογία βιώσιμων μελετών, ε, βιώσιμης μελέτης επιπτώσεων, βιώσιμης αξιολόγησης επιπτώσεων ε, και επίσης προτάσεις για τις διαβουλεύσεις των ελευθέρων ελευθέρων, ε, ζωνών ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών και ε, επίσης για τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε με την Κορέα. Ε, η Κομισιόν έχει επίσης δηλώσει τις προθέσεις της για ε, βάση του ψηφίσματος των κοινωνικών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια των ε, εργασιακών συμβάσεων. Αυτό, αυτή η πρόταση για την εξωτερική διάσταση, ε, διάσταση κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών πιστεύω ότι θα προωθήσει το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα και είναι μάλιστα και πολύ επίκαιρη η, έκθεση, η πρόταση αυτή σχετικά με τα θέματα τα οποία συζητάτε, συζη, συζητείτε εσείς και αναφέρονται στο ψήφισμα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ το θέμα της εταιρική ευθύνης βεβαίως ε, ε, είναι και αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική αυτή η εταιρική ευθύνη το έχουμε συζητήσει στο Κοινοβούλιο στο παρελθόν και η Κομισιόν 16 Φεβρουαρίου προθεσμία τροπολογιών για την γνωμοδότηση του κυρίου Φάμπρ ε, έχετε τελικά σχόλια κύριε Σιγητά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι ε, διατύπωσαν θερμά λόγια για, για το ταπεινό μου άτομο. Ο παλιός μου φίλος ο Αλεχάνδρο Θέρκας. Τόσα χρόνια που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπω συνέχεια τις προσπάθειες να καταληθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό υπόδειγμα στο οποίο βασίζεται η, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Για τον κύριο Κοφεράτη. Θέλω να τον ευχαριστήσω επίσης για τα λόγια και τα ενδιαφέροντα σχόλια που έκανα και στην Κομισιόν. Θέλω να πω ότι είναι καιρός να δημοσιεύσει αυτά τα οποία μέχρι στιγμή είναι εμπιστευτικά στη συμφωνία με την Ινδία όπου υπάρχει ο κίνδυνος του κοινωνικού dumping. Σας ευχαριστώ και ελπίζω οι τροπολογίες που θα κατατεθούν να είναι όσο το λιγότερο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. 16 Φεβρουαρίου τροπολογίες, 13 Απριλίου στην Επιτροπή μας και τον Ιούνιο, αν θέλει ο Θεός, στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέντε θα κάνουμε τις ψηφοφορίες. Θα κάνουμε λοιπόν μια διακοπή μέχρι τις 5 παραπέντε αλλά θα ξεκινήσουμε οι ψηφοφορίες 5 ακριβώς. Θα αρχίσουμε την ψηφοφορία σε ένα λεπτό. Έχετε τις κάρτες σας μαζί, ελπίζω. Um, λοιπόν, αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπο... Για την... Επί της παραγράφου 1, τροπολογία 26 ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ κατά απορρίπτεται 8, 28 υπέρ κατά όχι η συμβιβαστική α δεκτή 28, 29, 30, 31 αποσύρονται. Η συμβαστική α εγκρίθηκε. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συνεβαστική β υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 51 καταπίπτει, 52, 53, 54 αποσύρονται, 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική C, γάμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αυτό σημαίνει 56 καταπίπτει, 57, 59 ε, αποσύρονται, 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή 65-66 αποσύρονται 67 68 69 απορρίπτεται 70-71 απορρίπτονται 71 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές Πρέπει να ελέγξουμε. 70 αποσύρεται, 71 ψηφίζεται ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 υπέρ 26 κατά. Απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 αποσύρεται 76 ψηφίζουμε 76 υπέρ κατά αποχές απο, απορρίπτεται συμβιβασμός ε συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 αποσύρεται 78 80 3, 14 καταπίπτει Α, ΙΜΚΟ 4, το τελευταίο μέρος ως προσθήκη της συμβαστικής ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται το ΙΜΚΟ 4. ΙΚΟΝ 2 εγκρίνεται χωρίς ψήφο, το ίδιο ΙΚΟΝ 9, ΙΚΟΝ 10 επίσης. Πάμε στο 82, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προχωράμε κάτω στο 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 είναι διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε, προχωρούμε στο 108, στην 108, όχι, 104. 104. 104. Ψηφίζουμε 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Όχι λάθος. 106 λέει η πρόεδρος. 106 πρέπει να ψηφιστεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχές την 107 ε, τι έγινε. Ναι, έχετε δίκιο. Η 107. Ζητείτε διαγραφή. 107 που ζητεί διαγραφή. Α, έχει αποσυρθεί. Α, έχει αποσυρθεί. Μόλις το πληροφορήθηκα. Ευχαριστώ. 108 την, ψηφίσαμε. Συμβιβαστική ε, H. Εκεί είμαστε. Ο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Αποχές δεκτή. Εκατόν Προχωρούμε στην 125. Υπέρ. 125. Υπέρ. Τώρα ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική γιώτα. Άι. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εποσύρεται 126, 27 καταπίπτει. Όλες τις παρακάτω αποσύρονται. 129, 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 100, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχ... κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 134. Α, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψηφοφορία. 17 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 έχει αποσυρθεί. 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 15, προφορική της εισηγήτριας. Ζήτησα ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο, το πρώτο τμήμα είμαι υπέρ, το, στο δεύτερο τμήμα είμαι κατά. Κατά. Λοιπόν, προφορική τροπολογία σε δύο τμήματα της εισηγήτριας. το πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα είναι ολόκληρη παράγραφος. Και μετά ήθελα να διαγραφεί μία πρόταση, η οποία δεν είναι σωστή. Αυτά, τα λέτε, αυτά λέει η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, στο πρώτο τμήμα να, να, παραμείνει και το δεύτερο να διαγραφεί. Αλλά δεν έχω το αγγλικό κείμενο μπροστά μου. If Αν θέλετε ξεχωριστή ψηφοφορία, εντάξει, λέει η πρόεδρος. Προφορική τροπολογία. Υπέρ του πρώτου τμήματος, ακατά, αποχές, δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ωραία. 109 έχει αποσύρθει. Συμβιβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα προχωράμε στην 149. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150. Υπέρ, κατά, αποχές. Πρέπει να το... Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. 150 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ε, έχουμε μία ψήφο παραπάνω του ΕΛΚ. Προσέξτε, παρακαλώ. Ακόμα έχουμε μία ψήφο πλεονάζει από το ΕΛΚ. Εντάξει, εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Πέρα τη ψηφοφορία 14 υπέρ 27 κατά απορρίπτεται. 27 κατά απορρίπτεται. 151 έχει υποσυρθεί. 152 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, προχωράμε προς τα κάτω ώρα καταπίπτουν μέχρι μέχρι την 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 ε, ζητά διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 έχει αποσυρθεί, 169 καταπίπτει, ε, όχι, όχι, δεν καταπίπτει. 169, ψηφίστε παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική L, λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Απορρίπτονται οι επόμενες. Προχωράμε Συμβαστική μη, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε στην οίκον 5. Πρέπει να ψηφίσουμε την Econ 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ήμκο 2, το τελευταίο τμήμα να ψηφιστεί υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 186 επεσήρθη. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική νη υπέρ κατά αποχές δεκτή. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 έχει υποσυρθεί Ξεχωριστή ψηφοφορία στην 191. Πρώτο τμήμα της 191 υπέρ Κατά. κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονικά την 192. Άρχεται η ψηφοφορία. Πώς ψηφίσατε. Έληξε ψηφοφορία. 25 υπέρ, 17 κατά, δεκτή. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωση. 195 ζητά διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 197-198 έχουν αποσυρθεί. Συμβαστική όμικρον υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Α, και 206 έχει περιληφθεί στη συμβαστική, αλλά δεν έχει αποσυρθεί, οπότε καταπίπτει. Προχωρούμε στην 207, η οποία μόλις απεσύρθη, ωραία, συμβιβαστική. Α, μόλις μας είπαν ότι έχει αποσυρθεί η 207 από τον συντάκτη. Ο συντάκτης τη 207 την απέσυρα. Ωραία. Συμβιβαστική π. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε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 Vote Πέρα τη ψηφοφορία. 27 υπέρ. 20 κατά. Δεκτή. 2-20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2-2-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 224 έχει αποσυρθεί, 225 πρέπει να ψηφίσουμε. Τη 225 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 230 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 232 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. πάμε στη 2.38, όχι έχει αποσυρθεί, 2.39, 2.39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 2.40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 2.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 2.42 υπέρ, κατά, αποχές, Παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. 2.42. Άρχεται η ψηφοφορία. Επέρας ε, της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 23 κατά, ε, δεκτή. 2.43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.47 έχει προσυρθεί 2.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ρο υπέρ κατά αποχές δεκτή 261. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266 ζητά διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται συμβιβαστική S, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Νομίζω και 280 και η 285 απεσύρθη, πάμε στο συνδυαστική ΤΑΦ, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 291, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 292, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική U, υπέρ. Κατά, αποχές, Δεκτή. Πάμε στην 300, 300 υπέρ. Κατά. Ξανά την 300 υπέρ. Δεν είχαμε ακόμα τελειώσει όταν ζητήσατε έλεγχο. Λοιπόν, 300 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 3-0-1, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές δεκτή Πάμε στην 310 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 311 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 313 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, όχι, νομίζω είναι σαφές. Νομίζω απορρίπτεται. Απορρίφθη. 315 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 316 ε, έχει αποσυρθεί. Α, την 3.15 παρακαλώ. 3.15 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. ψηφοφορίας. Υπέρ 19. Κατά 28 απορρίπτεται. 3.16 έχει αποσυρθεί. 3.17 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.18 ναι. υπέρ. Α, είναι προφορική τροπολογία να διαγραφεί η λέξη εκοφήν και να αντικαθεστεί. Ε, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 318. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τις 23 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. 3.19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οίκον υιοθετήθηκε χωρίς ψήφο όπως ε, όλες τις οίκονα από 26 μέχρι 28, 31, 30, 44, 40. Η συγγήτρια πει 44. Θα ήθελα να εξασφαλίσω την ε, συνοχή ε, στην ε, ψηφοφορία. Έχουμε βάλει τις τροπολογίες της οίκων σε διαφορετική, σε όχι αριθμητική σειρά, γιατί έτσι είναι πιο λογικό. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την περίεργη σειρά των τροπολογιών. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει η πρόεδρος. Όσον αφορά την αρρύθμιση μπορούμε να τα, να τα τσεκάρουμε αυτά αργότερα. 3.21 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 3.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ε, συμβαστική W υπέρ κατά αποχές δεκτή. προχωράμε στην 329 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 330 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 331 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 332 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 333 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.39 έχει αποσυρθεί. 3.40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3.41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα μπορούσαμε να πάρουμε όλες τις τροπολογίες από το 3.42 μέχρι το 3.50. Δεν θέλετε. Καλά, τότε ξεχωριστά καθεμή. Πού είμαστε. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.43 έχει υποσύρθει. 3.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, 346 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 347 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 348 υποσυρθεί, 349 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 350 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 352 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 354 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική χ, εξ, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 355, 355, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 356, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 357, ζητά διαγραφή μαζί με την 358. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 359, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 360, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 361, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 362, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Y, Y, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πάμε στην ΙΜΚΟ 16, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Νομίζω. Να ξαναψηφίσουμε την ΙΜΚΟ 16, υπέρ αποχές, ναι, οπωσδήποτε. Δεκτή. 366 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 367 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 368 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 369 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 370 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 371 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 372 ζητά διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 375 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ζήτα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε στη συμβαστική 2α. AA. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Προχωρούμε στην 390. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 391 και 392. 393, 395 ζητούν διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 3-9-4-3-9-6 απεσύρθη, 3-9-7 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. κατά, ΒΒ υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τετρακόσια δύο. Τετρακόσια δύο υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική CC υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4.11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4.12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4.13 υπέρ. Μαζί με την 4.14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική DD, δέλτα δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, α, απορρί, ε, συγγνώμη, ε, δεκτή, λέει ο πρόεδρος. Έχω τρελαθεί, λέει εδώ. Συμβαστική DD πέρασε. Δεκτή. Ήμκο 24, Ήμκο 24, υπέρ, κατά, αποχές, Παρακαλώ ηλεκτρονικά την ΙΜΚΟ 24. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. ΙΜΚΟ 24. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. 416 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 417 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οίκον 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε ε υπέρ κατά Αποχέ. Δεκτεί. 423. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 424. Υπέρ. Κατά. Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 424. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, είναι σαφές λέει η πρόεδρος. 4.24. 424, λέει η πρόεδρος τροπολογία. 424 που ζητάει διαγραφή. Πέραση ψηφοφορίας 44 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, δεκτή. Τώρα, πάμε στην 428, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτε 429, υπέρ, κατά. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά την 429, άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι έχουμε μία παραπάνω ψήφο από το ΕΛΚ. Α, εντάξει, διορθώθηκε. Πέρα στις ψηφοφορίες για την 429. 18 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. Πάμε στην εικόν στις Οίκον 35-49. Πάμε στην Οίκον 45 που πρέπει να ψηφιστεί. Οίκον 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οίκον 47 χωρίς ψήφο. 48 χωρίς ψήφο. Οίκον 24. Προφορική τροπολογία. Οίκον 24 μετά από τις λέξεις ε, να προστατεύσει, να προσθέσουμε το, το απόθεμα, το book reserve. Λοιπόν, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Η 45 απερίφθη λέει η συγγήτρια. Ωραία, ωραία. Η 45 ε, πράγματι λέει η πρόεδρος απερίφθη έχουμε προχωρήσει τώρα στην οίκον 24 με την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή. 4.31-4.33 ταυτόσημες. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 4... 32 έχει αποσυρθεί. Ε, συμβαστική FF υπέρ, κατά, Αποχές. Δεκτή. Προχωράμε και ψηφίζουμε το μεσαίο τμήμα της 439. Μόνο το μεσαίο τμήμα, middle part, του 439. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4.40 ζητά διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική G. G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4-4-3. Α. Mm. 4-4-3. Υπέρ. Δύσκολα συγγήτρια. Εάν έχω, αν το κατάλαβα σωστά, ψηφίσαμε μια συμβιβαστική. Α, λάθος λέει η συγγήτρια. Η 4-4-2 καταπίπτει, διότι ψηφίσαμε το, το την προηγούμενη συμβιβαστική, το συμβιβασμό HH. 4-4-3 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, συμβιβαστική HH, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πάμε στην 451 υπέρ, κα, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 452 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 453 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβασμό, συμβαστική 2 2-Ι-Ι. αι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οίκον 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οίκον 56 μόνο το τελευταίο τμήμα. Οίκον το 56 τελευταίο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 4-5-8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-60-4-61 έχουν αποσυρθεί 4-62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκτιμώντας α Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 είναι συμβατή με την τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Το ίδιο ισχύει και για την 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 9 έχει υποσυρθεί 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 11 είναι συμβατή υπέρ κατά απερίφθη. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 έχει αποσυρθεί. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ, υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 15 άρχεται η ψηφοφορία νομίζω ότι μπορεί να έχει γίνει δεκτή Πέρας της ψηφοφορίας 26 υπέρ 18 κατά. Μία αποχή δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε την 16 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 29 υπέρ 18 κατά δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 έχει υποσυρθεί 20 υπέρ κατά απο... παρακαλώ ηλεκτρονικά την 20 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας 26 υπέρ 21 κατά δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 πρώτο τμήμα αποδεκτό δεύτερο τμήμα δεν είναι αποδεκτό ψηφίζουμε πρώτο τμήμα της 22 υπέρ κατά Παρακαλώ να ελέγξουμε την 22, πρώτο τμήμα, 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη της ψηφοφορίας, ναι, απερίφθη. 17 υπέρ 27 κατά απερίφθη. 23, 24, 25 όπως ήρθε. Οπότε προχωράμε στις τροπολογίες από το ΦΑΜ, ε, α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. C, ΦΑΜ, C, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. D, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή ε δεκτή, ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές δεκτή, F υπέρ κατά αποχές δεκτή, H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, J I υπέρ κατά αποχέ, αποχές απορρίπτεται, J υπέρ κατά αποχές δεκτή, K κάπα υπέρ ακαλύφθηκε από την F, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. L, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. M, μη, υπέρ, α, καλύπτεται από το φαμ α, α, It's It Καλύφθηκε ήδη από το ΑΦΑΜ, Α, F και H. Καλύφθηκε από, την πρώτη τροπολογία του, της ΦΑΜ, ΦΑΜ α Παρόλα όμως, παρόλα αυτά, Ας την ψηφίσουμε, λέει η πρόεδρος. Δεν θέλω να έχω επικαλύψεις, λέει η συγγήτρια. Κύριε Στέρξ, πρέπει να ψηφίσουμε γιατί η Α απερίφθη. Ένα λεπτό λέει η πρόεδρος. Η ΦΑΜ Α απερίφθη. Καλύπτεται όμως από το H και το F. Η ναι. F έγινε δεκτή. Ναι, λέει πρόεδρος, αλλά θα καλυπτόταν μόνο εάν είχε γίνει δεκτή η ΦΑΜ Α, η οποία δεν έγινε δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, απερίφθη. ΦΑΜ Ωμικρόν η προηγούμενη απερίφθη και η νη και η όμικρον απερίφθησαν. Παύλε, citations, ένα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, δύο και 3 αποσύρθηκαν, τέσσερα, προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, φαμ, παύλα ένα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, φαμ, παύλα, 2, ε, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 118 προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. κάποια, κάποια ψήφος λείπει. Κάποιος λείπει. Α, εντάξει, όλα είναι εντάξει. Έληξε η ψηφοφορία. 40 υπέρ. 6 κατά. Μία αποχή. Συγχαίρω την εισηγήτρια, την κυρία Όπεν Ρόιτεν. Ακολουθεί τώρα η... μια στιγμή η κυρία Ρόιτεν. Θέλω να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω, ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη, αλλά ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πάμε κατευθείαν στην ε, γνωμοδότηση του κύριου Κοφεράτη για τις μελλοντικέ συνέργειες που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μεταξύ του περιφερειακού και άλλων διαφορετικών ταμείων. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω χέρια. Μπορούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν να φύγουν το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην έκθεση του κ. Κομφεράτη. Υπέρ είπα. Κατά. Αποχές δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Συμβαστική α ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίντ. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Κάποιοι δεν τα χέρια τους. Έλεγχος ηλεκτρονικός τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 12. περασε 27 27-17 εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ. Is there any objection to an oral amendment on... Έχετε πρόβλημα με την προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 15, όχι. όχι. Κύριε Κομφεράτη, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία γιατί η προφορική τροποποίηση θα αλλάξει την 15. Πριν από την 15 πρέπει να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του κ. Ουγγουρεάνου. Ναι. Πρέπει να μας διευκρινίσετε για την ε, προφορική τροπολογία επειδή δεν βρίσκεται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Κύριε Κονφεράτη ή ο συντάκτης να μας εξηγήσει περί πρόκειται. Μπορείτε να μας πείτε τι λέει η προφορική τροπολογία. Τι λέει. Τι Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αλλάζει τις πολιτικές σε πολιτική. Και θέλει να διαγράψει τις δύο τελευταίες λέξεις. Από την έμφαση μέχρι την ανταγωνιστική συμπεριφορά. Κύριε Κοφεράτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέει ο κύριος Κοφεράτη. Ε, εντάξει. Ψηφίζουμε την προφορική, τη 15 με την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά. Αποχέ, δεκτή. Συμβαστική D, υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτή. 21 με προφορική τροποποίηση από τον συγητή που είναι μέσα στα χαρτιά σας. Ψήφι υπέρ 21. Κατά. Εποχές. <clears throat> Δεκτή. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 26. Ψήφι, ε, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία στην 26, σας είπα. Πέρας. Πλεονάζει ένας <clears throat> από το ΕΛΚ. Εντάξει, πέρας ψηφοφορίες για την 26. Ε, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 26-15-3. 27 ψήφι υπέρ κατά άποχες Εγκρίντ. 28 ψήφι υπέρ Για την 28 θέλετε να πείτε κάτι κύριε Ντόιτς. Θέλω την αποσύρω κύριε Πρόεδρε. Αποσύρεται 28. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση για τη συμβαστική F, σίγμα Ο λόγος στον κύριο Κοφεράτη, αν θέλει να πει κάτι για αυτή την προφορική τροπολογία. Έχετε το λόγο. Η τροποποίηση σε σχέση με το αρχικό κείμενο αφορά το τελικό κομμάτι. όπου αναφέρεται το θέμα της αύξησης σε υποθετικό επίπεδο του κοινωνικού ε, ταμείου εάν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο τροποποιεί το αρχικό κείμενο. Αν υπάρχει ανάγκη. Αν τηρήσεις, όχι, ψηφίζουμε συμβαστική F ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά έλεγχος για 34 ηλεκτρονικός άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 25-20 εγκρίνεται. Συγγνώμη, συμβαστική G. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 ψήφι πέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 39. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται 28-17. Τροπολογία 40. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 46-0 ομόφωνη έγκριση χωρίς αποχές, χωρίς αντιδρασπίπους. Συγχαρητήρια στον κύριο Κοφεράτη. Τώρα περνάμε σε διάφορες ψηφοφορίες για το γενικό προϋπολογισμό πρώτον για την απαλλαγή ως προς την Επιτροπή Τμήμα 3. Υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία, τον ίδιο εισηγητή, για την ανάπτυξη επαγγελματική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ, κατά, χε, εγκρίνεται. δύο Τροπολογία δύο Υπέρ, κατά, χε, εγκρίνεται. τρία Υπέρ, κατά, χε, εγκρίνεται. ηλεκτρονική επαλήθευση για τη γνωμοδότηση αυτή. Έληξε. 45-0 μία αποχή. Τώρα για το ίδρυμα βελτίου συνδικών διαβίωσης και εργασίας μία τροπολογία υπέρ. Τα. Επαλήθευση της τροπολογίας αυτής 1. Έληξε. 31-15-0. Εγκρίνεται. Ε, τώρα ηλεκτρονικά για το σχέδιο γνωμοδότηση στο σύνολό του άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 46 υπέρ 0 κατά 0 αποχές. Τώρα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφαλή και την Υγεία στην Εργασία. Μία τροπολογία πάλι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά ξανά για το σύνολο της γνωμοδότησης. Έληξε. 45 υπέρ, μία ψήφος κατά Επόμενο, Ευρωπαϊκό Ιδρύμα Επαγγελματική Εκπαίδευση. Δύο τροπολογίες. Η πρώτη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο. Έλξε. 45 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έληξαν οι ψηφοφορίε εδώ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στο Στρασβούργο, στι 14 Φεβρουαρίου, Στι 7 το απόγευμα. 14 Φεβρουαρίου είπα, στι 7 το απόγευμα. Χαίρετε. Ah.